Θα ξαναρχίσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά για μια γεμάτη σε διάταξη. Έχουμε την κατάσταση των Βεδοίδων στην Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Είναι αλήθεια ότι η σύγκρουση Ισραηλινών Παλαιστινίων Μα κάνει να παραβλέπουμε καμιά φορά τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Βεδουίνοι στο Ισραήλ. Μιλάμε για ένα πληθυσμό 140.000 Βεδουίνων Ντενεγεφ στο νότο του Ισραήλ, 12% του αραβικού πληθυσμού του Ισραήλ, που μέχρι τώρα έχει ξεχαστεί τελείως. Οι μισοί μένουν σε στρατόπεδα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος και που συνεχώς απειλούνται από κατεδάφιση. Έχουν επίσης καταστραφεί και υποδομές και υποδομές που έχει δημιουργήσει μάλιστα και η Γενική Διεύθυνση Κομισιόν. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι εδώ, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση των παιδιών στην ε, Μέση Ανατολή. Έχουμε καλέσει σήμερα εκπροσώπους υψηλής ποιότητας ο κ. Σαμπενάβη από το Πανεπιστήμιο Μπενκουριών του Ισραήλ πρώτα. Έχετε το λόγο για 8 λεπτά παρακαλώ. Okay, good morning everybody. I am really very pleased to be Καλημέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Ξέρω ότι έχω μόνο 8 λεπτά, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και ερωτήσεις. Είμαι ο Αλιάνα Κενάου, είναι, είμαι ε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπεν Χουριών και πριν από ένα μήνα ήμουν πρόεδρος ε, του Ακαδημαϊκού Κολεγίου του Αμπχάκρα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά κολεγία στο Ισραήλ. Ξεκίνησα ως ερευνητής είμαι πολύ αφοσιωμένος σε αυτό και λίγο πολιτική, αλλά κυρίως θέλω να επικεντρωθώ στην έρευνα. Εδώ και πολλά χρόνια λοιπόν κάνω έρευνα. Και ένα από το βασικό κομμάτι της έρευνάς μου, ερευνά τις επιπτώσεις της μετάβασης, οικονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτικές, ε, κοινωνικές που ε, πέρασαν στην κοινότητα των Βεδουίων. Ζω στο Ραχάτ, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, πόλεις των Βεδουίνων στο Ισραήλ. Ποτέ δεν μετακόμισα Πηγαίνω στον Καναδά που και που, μεν, αλλά ε, ποτέ δεν πήγα στο Τελαβίβ ε, ή στην Πάχρα πουθενάλλου. Όταν μιλάμε για την κοινότητα των Βεδουίνων, δεν μιλάμε ε, για ένα διαφορετικό λαό, αλλά για ένα κομμάτι, μια εθνότητα που ζει στη Γαλιλαία και στην δική μας περιοχή είναι περίπου το 30% του πληθυσμού της Νέγκευ πολύ σημαντικό νούμερο. 60% αυτού του πληθυσμού είναι κάτω των 18 ετών. Δηλαδή είναι νεαρός πληθυσμός στην πόλη του Ράχατ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αραβική πόλη στο Ισραήλ. 60.000 άτομα σε καθημερινή βάση, δηλαδή 26.000 παιδιά ε, πηγαίνουν στο σχολείο και 60.000 άνθρωποι ε, είναι, ε, ανήκουν σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, το 50% ζουν σε ε, αναγνωρισμένα χωριά και το υπόλοιπο σε μη αναγνωρισμένο χωριά. Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του εβραϊκού και του βεδουίνικου τομέα ως προς τις υπηρεσίες. Δεν θέλω να πάρω το μέρος κάποιου, απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερες επενδύσεις, αρκετούς πόρους που έχουν δοθεί στην κοινότητα των Βεδουίνων, αλλά δεν αρκεί. Ξεκίνησε ε, αυτό ε, και είδαμε λιγότερους ε, άντρες ή γυναίκες να φεύγουν από το σχολείο. Είδαμε περισσότερες γυναίκες να πηγαίνουν στο Λύκειο. Ε, μια μεγάλη διαφορά στη ζωή των Βεδουίνων. Υπάρχει αυτό το χάσμα μεταξύ των Εβραίων και των Βεδουίνων όσον αφορά στη χρηματοδότηση, όμως τώρα αρχίζουν να έρχονται περισσότερα κονδύλια στην κοινωνία των Βεδουίνων ε, ως κάποιος που έχει ασχοληθεί και με την εβραϊκή και την ε, βεδουίνικη κοινότητα να πω ότι στο παρελθόν είχαμε μόνο δύο-τρεις φοιτητές στο πανεπιστήμιο που ήταν βεδουίνοι. Αυτό που βλέπω τώρα είναι διαφορετικό και ίσως να είναι και μια κριτική για το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της πόλης και της περιφέρειας και όταν μιλάω για την περιφέρεια, μιλάω ε, και για τους Εβραίους. Να σας πω κάτι φίλοι μου. Όταν πριν από ένα μήνα ήμουν ακόμα πρόεδρος του Ακαδημαϊκού ε, Κολεγίου, ε, μόνο το 20% ήταν μη Εβραίοι. Ε, το 80% ήταν Εβραίοι. Πήγαμε στο Κριάτ Μαλάχη και σε άλλα χωριά εκεί γύρω και έστελνα τους φοιτητές για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει. Υπάρχει τεράστιο χάσμα. Ακόμα και στο Ραχάτ τα σπίτια είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στο Ριάτ Μαλάχη. Πριν από δύο χρόνια, 42 γιατροί Βεδουίνοι πέρασαν τις εξετάσεις για την ειδικότητα οι περισσότεροι από αυτούς ε, μπήκαν ε, στο Ισραηλινό σύστημα υγείας και ήταν από την πόλη μου. Από το χωριό αυτό πόσοι, μηδέν. Μην με παρεξηγείτε, υπάρχει αυτό το χάσμα, αλλά υπάρχει και κάτι που συμβαίνει τώρα στο Ισραήλ. Ως προς τις επενδύσεις που δίνονται πλέον, είναι περισσότερες. Φυσικά υπάρχει αυτό το θέμα μιας κοινωνίας σε μετάβαση. Ως Βεδουίνος και περήφανος Βεδουίνος, γιατί είμαι πολύ περήφανος για την ταυτότητά μου ως μουσουλμάνος Βεδουίνος στο Ισραήλ, ε, στο παρελθόν ε, ε, μιλούσα πάρα πολύ για τα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα της κοινωνίας η πολυγαμία. Ακόμα υπάρχει το επίπεδο βίας. Το λέω αυτό στην τηλεόραση. μα ακούν οι Βεδουίνοι. Είμαι ερευνητή. Είμαι πανεπιστημιακός. Θέλω να ακουστούν φωνές που έχουν σιωπήσει. Το επίπεδο της βίας είναι θέμα. Τα τελευταία χρόνια πάνω από χίλια άτομα Άραβες σκοτώθηκαν από άλλους Άραβες και αυτό το λέω ξεκάθαρα στα ΜΜΕ το, του Ισραήλ. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα που πραγματικά επηρεάζουν την εξέλιξη της κοινωνίας μας. Είναι κομμάτι της μετάβασης. Δεν είναι εύκολο βέβαια να περάσουμε από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στον σύγχρονο. Αλλά γιατί το λέω αυτό, για να κατανοήσετε ότι η κατάστασή μας δεν είναι εύκολη. Κάποια προβλήματα όσον αφορά στη γη υπάρχουν επίσης, ε, θα τα πούμε αργότερα. Ε, βλέπω αυτό το χάσμα και το επικρίνω και από τις δύο πλευρές. Κάτι άλλο που θέλουμε να συμβεί στην Ισραηλινή κοινωνία είναι η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα. Εγώ ε, είμαι και Καναδός, όχι μόνο Ισραηλινός. Βλέπετε, μπορώ να, να προσφύγω και στον Καναδά όποτε θέλω. Τέλος πάντων, όταν είδα τι συνέβη στην Ευρώπη, στο Ισραήλ, της είπα στον Καναδά, κατανόησα ότι πρέπει να προωθήσουμε το θέμα της πολυπολιτισμικότητας. Υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο Ισραήλ και εμείς ως Άραβες, ως Βεδουίνοι, ως Εβραίοι πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καθένας έχει τις αντιλήψεις του, τις προκαταλήψεις του, τα στερεότυπά του. Όμως πρέπει να μιλάμε για την πολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα και δεν μιλάω μόνο για τις δύο κοινότητες, μιλάω και για το σεξουαλικό προσανατολισμό και την πολιτική ιδεολογία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια αύξηση στον αριθμό των φοιτητών στην κοινωνία των Βεδουίνων, για να επανέλθω στο σύστημα εκπαίδευσης, κάθε χρόνο βλέπουμε 5.000 μαθητές να ε, αποφυτούν από τα λύκεια. Και μόνο το μισό από αυτούς πηγαίνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Στο σύστημα το εκπαιδευτικό, στα πανεπιστήμια, στα κολέγια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει αυτό το χάσμα στη χρηματοδότηση. Κοιτάξτε όμως τι έγινε στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης δόθηκαν χρήματα σε καθηγητές για να υποστηρίξουν τους φοιτητές. Πολλά χρήματα που πηγαίνουν για τους μη Εβραίους φοιτητές και την υποστήριξή τους για να μπουν στο σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτά είναι από την κυβέρνηση. Είναι καλά πράγματα. Να δούμε όλη την εικόνα. Δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχει και μαύρο και άσπρο. Εγώ είμαι πανεπιστημιακός. Είμαι ερευνητής. Δεν χρειάζομαι τους πολιτικούς. Ε, βλέπω την εικόνα ως έχει. Δεν είναι ούτε μαύρο ούτε άσπρο. Πρέπει επίσης να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Ισραήλ. Δυστυχώς οι περισσότεροι, τουλάχιστον οι Άραβες στο Ισραήλ, δεν κάνουν αυτή την, αυτόν τον διαχωρισμό. Σε ένα λεπτό τελειώνω. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν. Όμως, το κράτος του Ισραήλ, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να συμβιώσουμε σε αυτό. Άραβες και Εβραίοι. Και εμείς ως πολίτες του Ισραήλ πρέπει να πιέζουμε την κυβέρνηση κάποιες φορές να αλλάζει την πολιτική της για να έχουμε καλύτερες συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή. Η κυρία Ράιουα Αμπριάβρια έχει τώρα το λόγο. Είναι από το κέντρο για την πράσπιση των, ε, των ε, πολιτικών δικαιωμάτων στο Ισραήλ και η ιδέα να έχουμε ακριβώς αυτή την ακρόαση για τα δικαιώματα των Βεδοίνων είναι από αυτό το κέντρο. Έχουμε πολλές ε, άλλες ε, παρουσιάσεις. Θα πρέπει να μιλήσουμε λιγότερο, λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για την νομική πτυχή αυτού του ζητήματος. Ε, και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο ε, έχω ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. 70.000 ε, Εβεδουίνοι ζουν στο βορειοανατολικό Νεκουίφ και ασχολούνται με τη γεωργία και την εκτροφή ζώνων. Μέχρι το 48 ε, είχε υπάρξει η εκτίμηση ότι καλλιεργούσαν 5.000 εκτάρια από την γη Ναγκεφ ε, και μετά το 1948 ανάμεσα σε 11.000 και 18.000 Βεδουίνοι παρέμειναν. Στο Νέγκεφ οι Βεδουίνοι είναι αναπόσπαστο μέρος της αραβοπαλαιστινιακής μειονότητας και ταιριάζουν στην ε, παραδοσιακή περιγραφή, δηλαδή δηλαδή έχουν μοναδικά πολιτιστικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, έχουν δική τους ε, οργάνωση και ε, ένα, ε, το νέο σύγχρονο κράτος απειλεί την ταυτότητά τους δεν έχει, ε, πριν από λίγα χρόνια αναγνωρίστηκε ως αυτόχθονος ε, πληθυσμός. 46 ε, περίπου χωριά. Το κράτος του Ισραήλ αρνείται να τα αναγνωρίσει, να τα συμπεριλάβει στο χωροταξικό του σχεδιασμό. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των χωριών υπήρχαν προτού ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ το 1950 έγινε υποχρεωτική επανεγκατάσταση των Βεδουίνων σε ένα μικρότερο ε, χώρο, σε Σιάζ όπως ονομάζεται, δηλαδή σε ένα περιορισμένο χώρο. όλοι οι ε, οι Βεδουίνοι είχαν περιορισμούς ε, μετακίνησης και περιορισμούς σε σχέση με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούσαν να γυρίσουν στη γη τους και ζουν ως εσωτερικά εκτοπισμένοι εδώ και ε, πάνω από 60 χρόνια. Ακόμη και στη ζώνη Σιάτζ, οι Βεδουίνοι που εξακολουθούν να είναι εκεί δεν έχουν αναγνωρισμένους τίτλους ιδιοκτησίας από το κράτος του Ισραήλ. Ε, η έξωση και ο εκτοπισμός και η μετεγκατάσταση των Βεδουίνων ε, στο Νέγκεφ ε, ανάγκασε τους Βεδουίνους να εγκαταλείψουν την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής τους και την παραδοσιακή οικονομία που βασιζόταν σε εκτροφή και στην καλλιέργεια της γης. Όλη η γη δόθηκε σε Ισραηλινούς, <coughs> μεταφέρθηκαν στα κιμπουτσίμ και στις ε, τοπικούς, ε, ε, στοπικές τοπικές ενώσεις γεωργών. 30% ε, περίπου του Νεγκουίφ, περίπου 3 εκατομμύρια εκτάρια, αντιστοιχεί σε αυτή την υποχρεωτική μετεγκατάσταση ε, και ε, υπάρχουν 46 με αναγνωρισμένα χωριά Βεδουίνων αυτή τη στιγμή και μόνο 10 τώρα είναι να αναγνωριστούν και 35 δεν έχουν αναγνωριστεί και δεν εντάσσονται, όπως είπα, στο χωροταξικό σχεδιασμό. Για το Βόρειο Νεγκέφ, ε, βάσει της νομοθεσίας ε, του 65 για το χωροταξικό σχεδιασμό, ε, αγνοείται πλήρως και η η γη τους χαρακτηρίστηκε ως γεωργική γη σε άλλες κατηγορίες όπως βιομηχανική γη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι ότι απαγορεύτηκαν οι οικισμοί. Ως αποτέλεσμα, οι Βεδουίνοι ήταν σε μια ανυπόφορη κατάσταση που διαρκεί ακόμη. Νομικώς δεν μπορούν να έχουν άδεια κατασκευαστική και τα σπίτια στα οποία έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει και όπου έχουν μεγαλώσει οι οικογένειές τους θεωρούνται ε, εκτός σχεδίου ε, και απειλούνται με κατεδάφιση και με πρόστιμα. Ε, χίλια σπίτια περίπου κατεδαφίζονται το χρόνο ε, και φυσικά δεν είναι αγνωσμένα τα χωριά και δεν υπάρχει ε, κατασκευαστική άδεια, αλλά όχι επειδή θέλουν να παραβιάζουν νομοθεσία, αλλά επειδή είναι αναγκασμένοι, αναγκασμένοι λόγω της κρατικής πολιτικής που δεν αναγνωρίζει τη γη των Βεδουίνων. Πάνω από 100 φορές έχουν κατεδαφίσει ένα συγκεκριμένο χωριό, παραδείγματο χάρη. Οι κάτοικοι αυτών των χωριών σε μεγάλο βαθμό είναι οι αόρατοι πολίτες. Δεν έχουν ούτε βασικά δικαιώματα. Δεν, ε, είναι, δεν συνδέονται με τις αποχετεύσεις, ε, την ηλεκτροδότηση, την ίδρυυση, για να μην μιλήσω καν για ε, υπηρεσίες υγείας και παιδείας που είναι πολύ περιορισμένοι και να επαρκήσει η πρόσβαση. Και οι τίτλοι διεκτησίες φυσικά δεν αναγνωρίζονται. Δεν έχουν λοιπόν δικαίωμα σε βασικές υπηρεσίες και αυτή είναι μόνο μία έκφανση της συγκεντρωτικής πολιτικής του κράτους. Είναι με μέσω τιμωρίας και ένας μηχανισμός για να συνεχίσει να ασκεί την πίεση, ούτως ώστε να μεταφερθούν σε μία από τις 7 πόλεις που έχουν φτάσει, φτιάξει ειδικά για αυτούς. Ε, μέσα στο ΣΥΑΣ τους περιορίζουν ε, σε μία ιδιαίτερα μικρή ζώνη, αυτό είναι ο στόχο τη πολιτική, ούτω ώστε να εδραιωθεί ο πολιτικό έλεγχο των Βεδονίων και να ελαχιστοποιηθεί ε, το κόστος της υποδομής για την μετεγκατάσταση των οικισμών. Δεν αναγνωρίζει λοιπόν του οικισμούς και το Ισραήλ ε, ασκεί διακριτική μεταχείριση και συγκεντρωτική πολιτική κατά των κατοίκων αποκόπτοντας από την ζωή τους ε, στην Ήπεθρο και από τα γεωτεμάχια τους. Ε, ταυτόχρονα στον Έγκεφ πάνω από 100 εβραϊκοί οικισμοί υπάρχουν στη συνοικία Μπεστρέβα, μόνο 300 ε, κάτοικοι είναι και 16 διαφορετικά αγροκτήματα έχουν υποδομηθεί χωρίς άδεια και το κράτος αποφάσισε ε, αναδρομικά να αναγνωρίσει το καθεστώς και να τα εντάξει στο σχέδιο. Το Μάιο του 2015 το Ανώτερο Συμβουλίο αποφάσισε να εκενώσει το χωριό Ρεμχαλάν για να φτιάξει την Χεράν, μια Ισραηλινή πόλη. Ε, το χωροταξικό σχέδιο του ε, από τον Έχιο του Μπράουρ, από το Συμβούλιο Ασφαλείας, τελικά είχε ως στόχο μονομερός να εκτοπίσει τους Βεδουίνους και αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο πάνω από 70.000 Βεδουίνοι θα εκτοπιστούν εσωτερικά και ε, δεν μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της έξουσης οπότε ε, δεν ε, Υπάρχει καμία δυνατότητα διοικητική ε, διαδικασία ε, ε, για το ψήφισμα τώρα για την εγκατάσταση των οικισμών των Βεδουίνων. Σε μέσα σε μία πενταετία απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα και ένας Βεδουίνος ε, δεν έχει πρόσβαση έστω και για μία άδικη αποζημίωση ε, οποιασδήποτε αξιώσεις ε, ρυθμίζονται μέσα από αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα με την κατάσταση. Στα τέλη του 2013 το κράτος, παρότι έχει κρεμεί αυτό το σχέδιο, προχώρησε στον εκτοπισμό ε, περαιτέρω εκτοπισμό με άλλα ένδικα μέσα, μέσω του ε, χωροταξικού παραδείγματο χάρη νόμου ε, προς τον έγεφε Και οι Βεντουίνοι έχουν αποκοπεί από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και διαβίωσής τους. Δεν γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο μέσω διαφόρων διαφόρων δηλώσεων προβλέπεται η προστασία γενικότερα των ε, μειονοτήτων και ειδικότερα των αυτόχων ε, πληθυσμών. Ε, είναι συμβαλόμενο μέρο το Ισραήλ σε τέτοιε συμβάσει και πρέπει να του εξασφαλίσει κατάλληλη στέγη και διαφύλαξη της ταυτότητάς τους. Είναι ευπαθείς αυτή οι ομάδες, γι' αυτό δικαιούνται και προστασία βάσει του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, βάσει και τη δήλωση του ΟΗΕ για τους αυτόχρονους πληθυσμούς. Ε, συμπεριλαμβάνεται και υποχρέωση να μην υπάρχει με υποχρεωτική μετεγκατάσταση των αυτοχθόνων από τον ε, τόπο διαβίωσή του, χωρίς τη συνένεσή του και χωρί επαρκή ε, και δίκαιη αποζημίωση. Επίσης, οι αυτόχθονοι ε, πληθυσμοί διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα πάτρια εδάφη, του τους φυσικούς πόρους ε, και το κλωδόμημά τους και έχουν παραδοσιακά δικαίωμα ιδιοκτησίας και θα πρέπει να ανακτήσουν το γη και τα, τους πόρους που τους έχουν αφαιρεθεί αυθαίρετα. Εν κατακλείδη, ζητούμε από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο να καταθέσει ψήφισμα για την αναγνώριση των χωριών του Βεδένου στον Έγκεφ. 2. Να δημοσιεύει ανακοινοθέντα τύπου καταδικάζοντα δημόσια τι κατεδαφίσει και τη μη αναγνώριση των χωριών ε, Βεδουίνων. Τρίτον, ε, καλή τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισκεφθούν μια αναγνωρισμένα χωριά τέταρτον, ε, καλή την αντιπροσωπή για με το Ισραήλ να επισκεφθεί αυτά τα χωριά και να θέσει το ζήτημα ε, στις επαφές με την Κνεσέτ και στις, ε, με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει το θέμα των κατεδαφίσεων στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ και ε, στο Τελαβίβ ενθαρρύνουμε τον επικεφαλής την αντιπροσωπείας να επισκεφθεί το Ελχαρακή, το Ελχαράν και άλλα μια αναγνωσμένα χωριά πρωτού γίνουν κατεδαφίσεις σε πόρη για ευαισθητοποίηση και ανοικοδόμηση ε, σπιτιών ε, να χορηγηθεί η διεθνής προστασία στους Βεδοίνους και επίσης τον έγκυφ να επισκεφτείτε τα χωριά που έχουν ήδη κατεδαφιστεί. Πολύ σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ η κυρία Λένα Μανκούση Μαντέρη αξιωματικό σύνδεσμο από το Γραφείο για του Παλαιστινίου Πρόσφυγε. Ευχαριστούμε που με προσκαλέσατε. Όπω είπατε, εκπροσωπώ το Γραφείο του για τους Παλαιστινίου Πρόσφυγε στην Δυτική Όχθη, Λίβανο, Γάζα, Συρία. Θα σας μιλήσω για τη Δυτική Όχθη, όπου οι περισσότερες φυλές Βεδοίνων προήλθαν από την έρημο στο νότο του Ισραήλ. Έχουμε εντοπίσει πέντε κυρίως φυλές στην Δυτική Όχθη. Ατζαχαλίν, Αμπράμνε, Αρμετίν, Αλσάιτεν και Αλάσμε που περιλαμβάνουν πολλές κοινότητες στην Δυτική Όχθη, νότια της ε, Χευρώνας και αλλού. Εμφανίστηκαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας 40 και του 50 μετά από συγκρούσεις με τις ε, στρατικές δυνάμεις του Ισραήλ. Μετά τις εξελίξεις στις αρχές του 90, οι περισσότερες από αυτές τις κοινότητες πήγαν σε περιοχές που είναι υποκατοχή του Ισραήλ με πολύ περιοριστικούς όρους, ε, αστικούς ε, κλπ. Πολλές από αυτές τις περιοχές χρησιμοποιούνται στρατιωτικά από το Ισραήλ, αλλά κυρίως γύρω από την περιοχή της Ιερουσαλήμ έχουμε περιοχές οι οποίες προορίζονται για νέες εγκαταστάσεις. Έχουμε την περιοχή ε1 η οποία θα επιβάλλει την δημιουργία, μάλλον την μετακατάσταση 15.000 οικειών. Αυτό το βλέπουμε ως φαινόμενο αρκετά έντονα γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ και έτσι δημιουργείται ένας διάδρομος Δυτικής Όχθης και ε, Ανατολικής Ιερουσαλήμ και Ιερουσαλήμ γενικότερα και αυτό βεβαίως υποβαθμίζει και πλήττει το ενδεχόμενο δημιουργίας ε, δύο κρατών. Οι Ισραηλινές αρχές ενθαρρύνουν την εγκατάσταση επίκων και έχουν ε, εκτοπίσει αρκετές από αυτέ τι κοινότητε ε, Βεδουίνων, τι οποίε θεωρούν ω ε, εμπόδιο για αυτά τα επεκτατικά του σχέδια. Υπάρχουν λοιπόν αυτέ οι κοινότητε Βεδουίνων που μένουν και στην περιοχή Γ, στην Δυτική Όχθη, και οι οποίε αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μετακατάστασης ή εκτοπισμού από τι Ισραηλινέ αρχέ, κυρίω τι στρατιωτικέ αρχέ του Ισραήλ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω στις 7.500 η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι πρόσφυγες και καλύπτονται από την υπηρεσία που εκπροσωπώ εδώ. Έχουμε πάνω από 20 κοινότητες με 2.300 Βεδοινούς βρίσκονται στο διάδρομο Ιερουσαλήμ-Ιεριχώ και αυτοί βεβαίως αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο άμεσο εκτοπισμού. κοινότητες λοιπόν των Βεδουίνων υπόκεινται σε αυτό το καταπιωστικό περιβάλλον μέσω δράσεων του Ισραηλινού στρατού και της Ισραηλινής διοίκησης. Υποβάλλονται λοιπόν σε αυτό το μεγάλο κίνδυνο εκτοπισμού ως αποτέλεσμα αυτής της ε, καταστολής και βεβαίως παραβιάζοντας την ε, συνθήκη της Γενέβης. Την ενώ με καταπιστικό περιβάλλον. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι καταρχάς το ότι υπάρχουν μεγάλοι περιορισμοί όσον αφορά το αστικό περιβάλλον. Τα σχέδια, τα χωροτακτικά, τα οποία υποβάλλονται πρέπει να υποβληθούν στις ε, Ισραηλινές αρχές για υποδομές, βασικές υπηρεσίες, ε, κοινοφελή, ε, σχέδια κτλ. Όλα αυτά τα προγράμματα και τα σχέδια και αιτήσει απορρίπτονται συστηματικά οι κοινότητες αντιμετωπίζουν και ένα συνεχό κίνδυνο κατεδαφίσεων των υποδομών τους και συνεχούς εκτοπισμού. Έχουμε εκφοβισμούς από τις Ισραηλινές αρχές, κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά επίσης. Καθώς στρατιώτες αλλά και άλλοι εισέρχονται σε αυτές τις ε, κοινότητες, ε, βγάζουν φωτογραφίες, απειλούν και τους αθαρρύνουν να δεχτούν τις προσφορές μετεγκατάστασης. Υπάρχει απόρριψη της πρόσβασης στην γη, κάτι το οποίο βεβαίως υποβαθμίζει τις δυνατότητες επιβίωσης αυτών των κοινοτήτων. Και βεβαίως είχαμε και επεισόδια βίας και εκφοβισμού, το οποίο και αυτό βεβαίως υποστηρίζει αυτό το καταπιστικό περιβάλλον το οποίο σας περιγράφω. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια βίας γίνονται όλο και πιο συχνά. Είναι σχετικά σύμφω, πρόσφατο συγγνώμη, φαινόμενο με τρόπο οργανωμένο, αλλά ακολουθεί βεβαίω και την εξέλιξη της Ισραηλινής πολιτικής. Οι υπουργοί, αρκετοί υπουργοί του Ισραήλ και αξιωματούχοι διαμένουν σε αυτές τις περιοχές ως ε, έπικοι. Και μάλιστα και ο ο πρεσβευτή του ΟΗΕ δέχτηκε αυτό επίθεση στα πλαίσια της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Προσπαθούν λοιπόν να εκτοπίσουν τις κοινότητε Βεδοίνων οι Ισραηλινές αρχές. Τώρα, σε σχέση με αυτού τους Βεδοίνους που αποδέχτηκαν την μεταφορά αυτή ή τους υποχρέωσαν και στις δύο περιπτώσεις το θεωρούμε ως καταπιστικό περιβάλλον και καταναγκαστική αποχώρηση αυτών των βεδοίνων. Και αν αυτό αποδειχθεί ως φαινόμενο επαναλαμβανόμενο, τότε αυτό αποτελεί βέβαια κατάφορη παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης. Έχουμε επίσης και άλλες παράνομες δράσεις, όπως η, η οικοδόμηση επιπλέον οικειών επίκων σε κατεχόμενα εδάφη. Έχουμε λοιπόν συνεχείς παράνομες πράξεις εκ μέρους των Ισραηλινών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουν στη διεθνή κοινότητα ότι έχουν εκφράσει οι Βεδοίνοι την αντίθεσή τους σε αυτή την μετεκατάσταση, σε αυτή τη μεταφορά σε άλλα μέρη, γιατί βεβαίως ε, με αυτόν τον τρόπο θα καταστραφεί ο κοινωνικός του ιστός, ο, ο τρόπος ζωής τους κλπ. Οι Βεδουίνοι θέλουν βεβαίως να παραμείνουν στα εδάφη τους και ζητούν βεβαίως και λύσεις όσον αφορά τα θέματα χωροταξίας και αστικού σχεδιασμού. Το Ισραήλ ως ε, δύναμη κατοχής έχει υπό το διεθνέ καθεστώ αρκετέ υποχρεώσει και υπό το ανθρωπιστικό καθεστώ. Αυτέ οι υποχρεώσει αφορούν βεβαίω την προστασία του πληθυσμού που προστατεύεται υπό τη συνθήκη τη Γενέβη επειδή διαμένει στα εδάφη τα οποία κατέχει το Ισραήλ ω δύναμη κατοχή. και αυτή η προστασία αναφέρεται στο 49 άρθρο τη συνθήκη και διασφαλίζει το και λέει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να αποτρέπει οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, θα πρέπει να προστατεύει την ε, περιουσία των τοπικών κοινοτήτων και θα πρέπει βεβαίως να μην επιτρέπει την καταστροφή των υποδομών αυτών των κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίνει βεβαίως και την, τα βασικά, τις βασικές υπηρεσίες υγιεινής ε, και κοινοφιλών υπηρεσιών. Όλα αυτά λοιπόν δυστυχώς μας δείχνουν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται όσον αφορά τη μετακατάσταση αυτών των κοινοτήτων Βεδουίνων. Πάντως αυτό το καταπιστικό πλαίσιο που σας περιέγραψα για το οποίο οδηγεί στην απομάκρυση αυτών των κοινοτήτων. Το 60% των Παλαιστινίων Βεδουίνων είναι παιδιά και υποχρεούνται να μετεκατασταθούν μακριά σε, από εδάφη στα οποία κατοικούσαν εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια, ως δύναμη κατοχής, το Ισραήλ θα πρέπει να σέβεται την, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των οικογενειών. Πάντοτε σύμφωνα με την ε, συνθήκη της Γενέβης θα πρέπει να προστατεύονται και οι χώροι κατοικίας αυτών των ατόμων και να μην υπάρχει παρέμβαση οποιασδήποτε σε αυτή. Τα τωρινά λοιπόν σχέδια μετεγκατάσταση προκαλούν σοβαρές ανησυχίες υπό το διεθνές δίκαιο και θα θέλαμε να, να, παραθέσουμε και την Γενικό του ΙΕ που είπε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μαζικές μετακαταστάσεις πληθυσμού εκτοπισμού στην ουσία που απαγορεύεται, κάτι το οποίο απαγορεύεται από τη συνθήκη της Γενέβης και από το Διεθνές των Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Καρίμ Γιουμπράν από την Νίκη Πετσελέμ.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 I Σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό ε, που σας ακούμε, ακούμε την ε, κατάσταση όπως την περιγράφετε και ε, θα εργαστούμε εδώ τόσο ώστε να διαδώσουμε αυτή τη μαρτυρία σας. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Να ξέρετε όλοι ότι συζητάμε το θέμα αυτό με την παρουσία εκπροσώπων των πρεσβειών Παλαιστίνης και Ισραήλ. Αν έχουμε χρόνο θα τους δώσουμε το λόγο, αλλά δύσκολο μου φαίνεται γιατί πρέπει να πάρουν το λόγο και οι συνάδελφοι οι ευρωβουλευτές. Ε, καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Παντσέρη. Να σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι γιατί ξέρετε ότι στις 11 και 4 θα πρέπει να διακόψουμε για να πάμε στη συζήτηση στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με τον Επίτροπο Χάν. Κύριε Παντσέρη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας και συμφωνώ βέβαια. Νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά εδώ να επαναλάβουμε την φράση του Αμοσός για τη σύγκρουση. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αγώνα του καλού κατά του κακού, αλλά κατά του δικαίου, του κατά του αδίκου. Γιατί έχει ξεκάθαρα άδικο εδώ το Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν αυτό το καταπιστικό περιβάλλον, έχουμε τους εκτοπισμούς των Βεδουίνων, έχουμε αυτές τις ε, τοποθεσίες οι οποίες είναι για μετακατάσταση αλλά είναι ακατάλληλες και ανθρωπιστικά. Κάποιες κοινότητες βρίσκονται σε περιοχές όπου έχουμε την επέκταση των Ισραηλινών επίκων και νομίζω ότι δεν έχουμε να κάνουμε με εκτοπισμούς κατά το οποίο απαγορεύεται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Δεν ερωτώνται αυτές οι κοινότητες και βρίσκονται σε μια θέση όπου δεν έχουν εναλλακτικέ. Και αυτό βεβαίω μεταφράζεται σε συνεχείς επαφές σε άτομα και σε υποδομές, συμπεριλαμβάνω και των υποδομών της Ένωσης εκ μέρους των επίκων, των Ισραηλινών, που δρούν σε καθώς πλήρους ατιμορρησίας. Κάνουν επιθέσεις σε σχολεία, σε εκνεοτροφικές υποδομές, σε υποδομές γενικότερα. Οπότε συμμερίζουμε απόλυτα αυτά που έλεγε η κυρία Αμποράβια προηγουμένως και θα ζητήσω εκ μέρους της ομάδας μας να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα κατεπήγων για τους εκτοπισμούς των Βεδοίνων στην επόμενη σύνοδο του Στρασβούργου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πανθέρη, κύριε Ροντρίγκες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη είπε ότι ήθελα και εγώ να πω. Δεν καταφέρνω να διαβάσω το όνομά σας, καθηγητά. Όταν μιλάτε για πολυφωνία και πολυπολιτισμική, πολυπολιτισμικό περιβάλλον, πολλές φορές υπάρχουν ε, αυτοί που ανέχονται τους άλλους ε, και αυτοί που γίνονται ανεκτοί. Ε, και μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση με την κατάσταση πριν από 10-15 χρόνια και θα ήθελα να παραθέσω ένα πανεπιστημιακό που είπε ότι το ΠΑΟΕΠΛΕΝ έχει μια εθνοτική διάσταση. Εσείς πώς ε, ερμηνεύετε αυτά που είπε. Ευχαριστούμε κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που ακούσαμε. Συμφωνώ Έχω όμω δύο ερωτήματα προς την εξωτερική υπηρεσία Εξωτερική δράσης. Τι κάνετε για τη κατεδάφιση των ε, προγραμμάτων που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σπίτια κατεδαφίζουν ε, τον Βεδουίνων ε, το Μάιο, το συζητήσαμε στην Ολομέλεια. Δεν έκανε τίποτα όμως κυρία Μαγκερίνη έκτοτε. Ε, παραμένουν οι απαθείς η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και επιτρέπει έτσι την κατεδάφιση. Αναφέρομαι σε ένα άρθρο από τις 7 Νοεμβρίου στον Ισραηλινό τύπο, όπου έλεγε ότι ε, η ομάδα εργασίας του Ισραηλινού Συμβουλίου αποφάσισε να ζητήσει αποζημίωση για τις ε, κατεδαφίσεις στη ζώνη ΣΥ και ε, για κύριε Μουσάβα, θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Είπατε ότι απειλούνται με κατεδάφιση των σπιτιών τους οι Βεδουίνοι. Θεωρείτε ότι οι διπλωμάτες έχουν, κάνουν αρκετά για να υπερασπιστούν ε, τους Βεδουινούς ή μόνο εμείς κινητοποιούμαστε. Ε, εγώ είμαι και στην αντιπροσωπεία και έχω, πάει, έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους. Τι άλλο μπορούν να κάνουν ε, οι διπλωμάτες, κατά τη γνώμη σας. Και, οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απειλούνται σοβαρά στο Ισραήλ. Πέρασε και ένα νομοσχέδιο για αυστηρότερα μέτρα. Εσείς μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας πλέον έτσι όπως έχουν οι περιορισμοί. Γιατί μας βοηθάτε και εσείς, εσείς μας τροφοδοτείτε με πληροφορίες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εμείς πρέπει να κινηθούμε, δικό μας ε, καθήκον και εμείς δεν κάνουμε αρκετά. Παροβιάζεται ε, η, νομοθεσία και δεν κάνουμε αρκετά. Ευχαριστούμε κύριο ε, Τσίπ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε περιγράψει μια κατάσταση των πραγμάτων όσα έχουν στις περιοχές που έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού Βεδουίνων. Ε, όπου και να βρίσκονται οι Βεδουίνοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι λόγω κουλτούρας και πολιτισμού είναι νομαδικός λαός. Όπου και αν βρίσκονται λοιπόν αντιμετωπίζουν προβλήματα που ε, οφείλονται στην κουλτούρα τους. Ε, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι πολύ φιλικός ως προς την κουλτούρα τους και αυτό ισχύει και για άλλους τομείς. Να ρωτήσω λοιπόν αν έχετε παρατηρήσει κάποια αποτελέσματα κατόπιν των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που έχετε διεξαγάγει. Πέρα από κάποια αρνητικά, έχετε δει να επιλύονται προβλήματα σε συγκεκριμένα μέρη. Υπάρχει κάποια θετική επίδραση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν επιληθεί δηλαδή προβλήματα που σχετίζονται με την κοινότητα των Βεδουίνων στην, ε, στην έρημο. Ναγκέφ, τι περιμένετε, ποια είναι τα στάδια, ε, ποια είναι τα βήματα, η δράση και η αντίδραση που περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο. Ο τελευταίος συνάδελφος, ο κύριος Γκερίνκα, έχει το λόγο. Έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να απαντήσουν και οι εισηγητές. Αν μιλάτε πολύ, θα μπορέσουν να απαντήσουν. Έχω ένα κεντρικό ερώτημα που είναι γιατί το Προεδρείο δεν κατάφερε ο εκπρόσωπος του Ισραήλ να είναι εδώ ως προσκεκλημένος. Υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Δεν είναι καλό να ακούμε μονομερείς απόψεις. Εδώ είναι. Αν ήσασταν εδώ, αν αφήνατε λίγο χρόνο θα μιλήσει. Το Ισραηλινό κράτος ε, πρέπει να φροντίζει όλη τη χώρα που δεν αποτελείται μόνο από φίλους. Πολλοί χιλιάδες ε, στο Ισραήλ εποφελούνται από την ελλειπή ε, νομική κατάσταση στο καθεστώς και το Ισραήλ λοιπόν θα έπρεπε να το ρωτήσουμε γιατί είναι έτσι η κατάσταση των Βεδουίνων. Γιατί ε, δεν κοιτάμε και τις άλλες χώρες της περιοχής. Ξέρουμε επίσης ότι εκατοντάδε. εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι ε, εκδιώκονται από τις αραβικές χώρες και πηγαίνουν στο Ισραήλ ως πρόσφυγες. Τους εκδιώκουν από τις πατρίδες τους Κύριε Γκερίκε. Δεν έχουμε χρόνο. Κάνουμε μια συζήτηση. Έχετε ερώτηση για τους συζητητές. Ξαναρωτάει ο Πρόεδρος. Γιατί πρέπει να απαντήσουν. Και πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις των βουλευτών. Αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτά που θα πούν οι άλλοι βουλευτές, μπορείτε να το κάνετε αργότερα. Αλλά για τα μέλη εδώ πέρα του πάνελ, τους συγητές, έχετε ερώτηση. Μπορείτε να συνεχίσετε αργότερα, αλλά πρώτα να απαντήσουν οι συγητές. Ωραία. Το ερώτημα. Ποια είναι η θέση τη Ισραηλινής πλευρά, Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Ωραία. Έχουμε καλέσει και την Ισραηλινή πλευρά. Δεν είναι όμω εδώ. όχι. Θα του δώσουμε το λόγο. Θα του δώσουμε το λόγο. Θα δώσω το λόγο πάντω ένα λεπτό στου προσκεκλημένου για να απαντήσουμε την ίδια σειρά με την οποία έλαβαν το λόγο. Παρακαλώ. No, Εσείς αρχίστε. Ευχαριστώ. Όταν ε, μιλούσα για αυτά τα χρόνια, γιατί ε, μιλούσα για τους Βεδουίνους στον Έγκεφ και στον Γκάλερ. Και υπάρχει χάσμα, όπως σας εξήγησα. Όποιος μελέτησε τις κατεδαφίσεις και πόσο επηρεάστηκαν τα παιδιά, ε, εγώ ήμουνα ο ίδιος, όχι ο Μπετσέλεμ, κανένας άλλος. Εγώ μίλησα στην κυβέρνηση και τους είπα τι κάνει αυτό στα παιδιά. Πολλά χρήματα έχουν διοχετευτεί για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Υπάρχουν περισσότεροι φοιτητές. Υπάρχει αλλαγή. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Δεν, χρειά, χρειάζεται, έχω τον τίτλο, δεν χρειάζεται να... Ε, την έδρα μου δεν χρειάζεται να... Δεν χρειάζομαι προαγωγή, δεν τα λέω αυτά γιατί χρειάζομαι κάτι. Υπάρχει σύγκρουση για τη γη και ε, θα πρέπει το Ισραηλινό κράτος με την κοινότητα των Βεδουίνων να λύσουν αυτό το πρόβλημα έγκαιρης ιδιοκτησίας. Υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να ρυθμιστεί. Για ταυτόχρονες πληθυσμούς παντού ανά τον κόσμο η πολυπληθυσμικότητα είναι βασική προϋπόθεση για να καταλάβουμε τους άλλους. Και εγώ τα τελευταία χρόνια αυτά που προσπαθώ να κάνω είναι να επηρεάσω το δημόσιο λόγο στο κράτος του Ισραήλ για να δεχτούν την ύπαρξη άλλων. Υπάρχει τεπελώριο χάσμα ανάμεσα στους Ισραηλινούς και στους Βεδουίνους, γιατί θεωρούν ότι είμαστε οι εχθροί. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα. Είναι στερεότυπα, είναι κλισέ, είναι ε, διακριτική μεταχείριση, δημιουργείται φόβος και αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε και για τις ερωτήσεις σας. Το βασικό είναι η ισορροπία δυνάμεων, η σχέση εξουσίας ανάμεσα σε, στους Ισραηλινούς που κυβερνούν και ε, τους Παλαιστινίους που είτε είναι Βεδουίνοι είτε πολίτες ε, του Παλαιστινιακού κράτους. Είναι διακριτική μεταχείριση και στόχος είναι η Παλαιστίνη. Δεν μπορεί να αυτό να κυρίσει η δημοκρατία του Ισραήλ. Γιατί είναι ε, δημοκρατικό και ελεύθερο το καθεστώς για τους Ισραηλούς και ανελεύθερο για τους Παλαιστινίους. Και κύριε, αν προσπαθείτε να κάνετε σύγκριση με ε, τη Μέση Ανατολή, να μην ήταν στο ε, νόση, αλλά αφού θέλει να ανήκει στις δυτικές χώρες, ε, στο δυτικό κλαμπ, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα επιθετικά μέσα για να κατεδαφίζει τα σπίτια των ανθρώπων. Τι θα κάνουν οι γυναίκες, τα παιδιά, οι άστεγοι μετά, μετά τις κατεδαφίσεις, δεν έχουν που να μείνουν. Είναι, είναι βασικά πράγματα που ζητάμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Σε αυτό το πάνελ ε, παρουσιάζουμε την, ε, παρουσιάσαμε την κατάσταση των βεβίνων που ζουν στο Ισραήλ. και είχαν γη εκεί. Εγώ στη δική μου παρουσίαση μίλησα για τη Δυτική Όχθη που είναι η υποκατοχή. Είναι σημαντικό. Πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται, να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτό προσπάθησα να το τονίσω ήδη στην παρουσίασή μου. Ζητούμε υποστήριξη πολιτική και οικονομική από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναγνωριστεί το καθεστώς τους, να μην χρειαστεί να φύγουν χάρη στη βοήθεια που θα μας δώσετε για να ασκήσουμε πίεση με τους, ε, τους εμπλεκόμενους φορείς για να πάψουν ε, αυτές οι διακριτικές μεταχειρίσεις. Πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και να έχουμε τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους τόσο ώστε οι ανθρωπιστικοί φορείς επιτόπου να μπορέσουν να ε, δραστηριοποιηθούν και να βοηθήσουν τους πάσχοντες. Ευχαριστούμε. Ακούσουμε τώρα την ε, εκπρόσωπο της ε, πρεσβείας του Ισραήλ για πολύ λίγο και μετά θα ακούσουμε την, τον εκπρόσωπο των Παλαιστινίων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι κάπως ανισόρροπη αυτή η παρουσίαση και διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα και έχει το στόχο μόνο πλέξη του Ισραήλ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεπής με την έλλειψη βούλησης για συντονισμό με τις Ισραηλινές αρχές όσον αφορά την δημιουργία υποδομών σε αυτή την περιοχή Γάμα. Όλα αυτά που είναι παράνομα, εκ νόμου θα πρέπει να φεύγουν. Οι Παλαιστίνοι έχουν δυνατότητες για προσφυγή στο Νότο Δικαστήριο και οι κατεδαφίσεις γίνονται τελικά μόνο με την έγκριση του ονοτάτου Δικαστηρίου. Όσον αφορά τώρα την Ένωση και τις χώρες που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός με την ΚΟΚΑΤ. Αν υπάρχει, έστω και αν υπάρχει διαφωνία για την ερμηνεία του ανθρωπιστικού δικαίου, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται την χώρα αυτή, το Ισραήλ. Στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν νομίζω να υπάρχουν παρενέργειε, συγγνώμη, παρερμηνίε του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Οπότε οι αποφάσει σε σχέση με την οικοδόμηση είναι νομικά δεσμευτικέ. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Καθηγητή, να πω ότι υπάρχει από δεκαετία του 70 μια υπηρεσία στο Υπουργείο Γεωργίας που ασχολείται ακριβώ με τα θέματα ιδιοκτησία των Βεδουίνων. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμό και συνεργασία στην περιοχή Γάμα με το Ισραήλ υπέρ των Παλαιστινίων για να αποφευχθούν ακριβώς μονομερείς ενέργειες οι οποίες οδηγούν στην επιδείνωση της κατάστασης για όλου. Ευχαριστώ. Να σας πω, λέει ο Πρόεδρος, ότι η ακρόασή μας έχει θέμα την κατάσταση των Βεδουίνων. Πάντως, να, να ακούσω την εκπρόσωπο της πρεσβείας του Ισραήλ να μιλά για ανισορροπία, η έλλειψη ισορροπίας, μου φαίνεται τουλάχιστον αστείο. Ο εκπρόσωπος της Παλαιστινικής Πρεσβείας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν προετοίμασα κάτι επίσημο. Να υπενθυμίσω μόνο στην εκπρόσωπο της δύναμης κατοχής για το ότι όταν μιλάμε για την περιοχή Γ, μιλάμε για περιοχή υποκατοχή κατά του διεθνούς δικαίου. Αυτό που μας εκπλήσει, Πρόεδρε, είναι αυτή η πολιτική μεταφοράς ε, πληθυσμών και καταστροφής ιδιοκτησιών περιουσιών Παλαιστινίων δεν είναι κάτι νέο. Από το 1948 ισχύει και εφαρμόζεται από το Ισραήλ και έχει ήδη τεκμηριωθεί ως πολιτική με συγκεκριμένα γεγονότα και τεκμήρια. Από το 67 και μετά έχει κατεδαφίσει 48.000 παλαιστινιακά σπίτια και υποδομές το Ισραήλ στα κατεχόμενα από το 67 μόνο. Και είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχουν 200, 230 περιοχές επίκων όπου έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου με τη μεταφορά αυτών των επίκων σε αυτές τις περιοχές και, τον, ε, και την εκδίωξη των Παλαιστινίων. Το δεύτερο που μας ε, σοκάρει, Προεδρία είναι το Ισραήλ. Είναι η μόνη χώρα που έχει ισχυρή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μιλάμε για γεγονότα που πηγαίνουν πίσω 60 χρόνια. Δεν μιλάμε για σημερινά μόνο γεγονότα. Και ξέρουμε ότι σε αυτές τις επικίες υπάρχουν και αξιωματούχοι Ισραηλινοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση και που συνεχίζουν να μην συνέβαινε τίποτα. Και πρόεδρε γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν και Ευρωπαίοι υπήκοοι με διπλή υπηκότητα από ευρωπαϊκές χώρες σε αυτούς τους χώρους επικισμού και οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει να είναι υπόλογοι για την παρουσία τους σε αυτούς τους χώρους επικισμού. Να σας ευχαριστήσω, λέει η Πρόεδρος. Δυστυχώς δεν είχαμε εκπρόσωπο από την ΕΙΑΔ επειδή αρρώστησε σήμερα το πρωί. Πάντως έχουμε ένα εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν από την ΕΚΟ. Μήπως θέλετε το λόγο. Έχει τελειώσει και ο χρόνος μας. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάντως για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των πρεσβειών Ισραήλ και Παλαιστίνης. Ευχαριστώ του προσκεκλημένους μα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να προασπίσουμε και να υπερασπιστούμε την κοινότητα των Βεδουίνων. Στο 1002 έχουμε τη συνάντηση με τον Επίτροπο Χάν.